Can we start? Μπορούμε να αρχίσουμε παρακαλώ. Um, good afternoon everybody. Can we start by... Καλησπέρα σε όλους Μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη ως ε, πρώτο θέμα. Καλώς πάρα πολύ γρήγορα μερικές ανακοινώσεις έχω να σας κάνω. Μεταδίδεται ζωντανά στο διαδίκτυο η συνεδρίασή μας και ορίζω οποιοδήποτε μας βλέπει, μας ακούει έξωθεν. Σας θυμίζω επίσης ότι έχουμε μια νέα έκδοση του newsletter το ενημερωτικού μας φιλανθείου. Έκανα ε, Πρέπει να σας πω ότι δέχτηκα σήμερα το πρωί ε, κάποια μέλη του ΚΟΡΕΠΕΡ, της Επιτροπής ε, Μονίμων Αντιπροσώπων και μας είπανε πόσο χρήσιμο τους ε, φαίνεται. Πραγματικά έχουν κάνει πολύ καλή οι εισηγητές, πολλή δουλειά και είναι πάρα πολύ καλό. Επίσης, έχω συναντηθεί αυτή την εβδομάδα με μέλη της Επιτροπής Κοινωνικής και Οικονομικής Επιτροπής, οι οποίοι θέλουν να εθαρρύνουν τους συζητητέ μας αν θέλουν να συνεργαστούν ε, με τα μέλη της ε, ΟΚΕ. Παρακαλώ να τους πλησιάσετε. Ε, έχουν και υποεπιτροπές και θέλουν να συνεργαστούν να φάκελο, με τους, με τους μας είναι η ηλεκτρονική επιτροπή, έχετε αυτή την εφαρμογή ε, και τα μέλη και η βοηθή και η πολιτική υπάλληλοι. Λοιπόν, είμαστε συνεδρίαση χωρίς ε, έγγραφα. Επίσης, θα έχουμε και κλεισμένο το θηρόν συνεδρία. Όχι, συγγνώμη. Από τη Γενική Διεύθυνση IPOL θα έρθει ένα τηλεοπτικό συνεργείο που θα τραβήξει μόνο εικόνες, όχι ήχο. Δεν ξέρω αυτό τι σημαίνει. Έχουμε βουβές συνεδριάσεις. Τι να πω. Μπορούμε να εγκρίνουμε τα πρακτικά ή να θεωρήσουμε ότι έχουν εγκριθεί αν δεν προβάλλει κανείς καμιά αντίρρηση. Αυτές ήταν ανακοινώσεις. Να σας ενημέρωσω για τις ε, διαπραγματεύσεις στο τριμερή διάλογο περιμένοντας να καταφτάσει ο Ανδρέας Σβάπ. Α, να τα αλλάξουμε και να πούμε πρώτα τα υπόλοιπα. Α, πριν αρχίσουμε ακόμα, σας έχει δοθεί ή θα σας δοθεί ένα σετ ε, εγγράφων που είναι ε, σύνοψη των δεσμεύσεων των επιτρόπων στο Κοινοβούλιο κατά την ακρόαση. Αυτά, ξέρετε, τα έχει παραγγείλει η αρμόδια Γενική Διεύθυνση. Δεν έχουμε την ευκαιρία να τα σχολιάσουμε. Απλώς αναφέρει τα όσα διεμήφθησαν ε, στις ακροάσεις και αν σε λίγα χρόνια δεν θέλουμε να ξανακούσουμε ολόκληρη την ακρόαση τρει ώρε. ε, χρειαζόμαστε ε, αυτά τα έγγραφα για να ανατρέξουμε. Ωραία, δεν αλλάζουμε τη μέση διάταξη αφού ήρθε ο κύριο Φαμπ να μα ενημερώσει ο ίδιο για τι διαπραγματεύσει μέχρι τώρα για το τριμερή διάλογο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Καθυστέρησα λέει ο κύριο Φαμπ στα αγγλικά και πρώτα πρέπει να ζητήσω συγγνώμη γι' αυτό. Είχαμε συνεδρίαση των σκιωδών για την οδηγία για την ασφάλεια των δικτύων και πρέπει να σας πω ότι εμείς επιμένουμε πάρα πολύ και εμένουμε στη γραμμή μας. Στις 14 Οκτωβρίου είχαμε ένα πρώτο άτυπο τριμερή διάλογο που ξεκίνησε παρόλο που δεν είχε καταφέρει να έχει επίσημη εντολή ακόμα η Ιταλική Προεδρία. Και παρακαλώ τους συναδέλφους τους Ιταλούς να απευθυνθούν και στην Ιταλική ε, Προεδρία για να επιταχύνει τα πράγματα, αλλά διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο έχουν νόημα εφόσον έχει και θέση το Συμβούλιο. Την Παρασκευή ελπίζω η Ιταλική Προεδρία να καταφέρει να αποσπάσει, να κερδίσει μια εντολή. Στις 11 Νοεμβρίου θα ξανασυνεδριάσουμε και γι' αυτό όπως είπαμε σήμερα το πρωί και επί τη βάση των σχεδόν εισηγητών στη συνεδρίαση αυτή είδα και την κυρία συνάδελφο Ντελ Καστίγιο, ε, και τον Φίλιπ Άλμπρεχτ από την Επιτροπή Ελευθεριών και τονίσαμε και πάλι ότι θέλουμε να επιτύχουμε το εξής. Η ασφάλεια ε, στο διαδίκτυο θα πρέπει να επικεντρωθεί σε κρίσιμες υποδομές και σε κάθε κράτη-μέλη θα πρέπει να προστατεύονται όλες οι υποδομές που αναφέρονται στο παράρτημα 2 της οδηγίας μετά την ψηφοφορία του Κοινοβουλίου και περιμένουμε από τα κράτη-μέλη, από το Συμβούλιο να δώσουν τουλάχιστον μια προοπτική για μια στρατηγική αλλά και επιχειρησιακή συνεργασία. Χωρίς μια τέτοια αξιόπιστη προοπτική δεν έχει κανένα νόημα η οδηγία. Γι' αυτό ελπίζουμε οι Ιταλοί ε, στο Συμβούλιο να καταφέρουν να πείσουν τους ομολόγους τους ότι είναι σημαντικό το βήμα που πρέπει να γίνει. Περισσότερα νομίζω δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή, εκτός του ότι ε, είμαι πάρα πολύ ευγνώμων στους σκιώδεις ηγητές για τη συνεισφορά τους. Okay, so is being... Ε, γίνεται λοιπόν κάποια πρόοδος από ό,τι φαίνεται. Αλλά από ό,τι φαίνεται το Συμβούλιο δεν έχει ακόμα την εντολή. Και ο εισηγητής και οι σκιώδεις κάνουν τη δουλειά τους και πολύ καλοί ε, προσπαθούν να πιέσουν το Συμβούλιο να αποκτήσει εντολή επιτέλους. Ε, παρακαλώ για την ΕΚΟ. Ευχαριστώ πολύ. Κατ' εξαίρεση θα μιλήσω αυτή τη φορά στα αγγλικά γιατί και οι σημειώσεις μου είναι στα αγγλικά. Θα ήθελα λοιπόν να σας μιλήσω για τις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του τρεμερούς διαλόγου. Στις 25 Σεπτεμβρίου λοιπόν αποφάσισε η ΙΜΚΟ να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή και το Συμβούλιο στο πλαίσιο τρεμερούς διαλόγου για να έχουμε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση για την πρόταση για το οικοσύστημα και είχαμε την εντολή μας με βάση την έκθεση που εγκρίναμε στην Επιτροπή και βάσει της οποίας εγκρίναμε και μία θέση στις 26 ε, Φεβρουαρίου σε πρώτη ανάγνωση. Η σύνθεση της διπραγματευτικής ομάδας ήταν η πρόεδρος Βίκη Φόρτ, υποφαινομένη ως εισηγήτρια, οι σκιώδεις εισηγητές και οι συντάκτες γνωμοδότησης των Επιτροπών ΛΥΠΕ και ΤΡΑΝ. Στις 8 Οκτωβρίου η διαπραγματευτική ομάδα του Κοινοβουλίου συναντήθηκε για να συμφωνήσει τη διαπραγματευτική εντολή. Την ίδια ημέρα το μεσημέρι έλαβαν χώρα οι πρώτες συναντήσεις, είχαμε τον πρώτο άτυπο του μερή διάλογο. Συζητήθηκαν κάποια πολιτικά ζητήματα, παραδείγματος χάρη η συνύπαρξη του e-call, το αν θα το ε, εντάξουμε και στις τεχνικές μονάδες, μονάδες υποστήριξη. αν θα πρέπει το e-call να είναι σωματωμένο ή όχι. Θέλαμε να δούμε την συμβατότητα με τις υπηρεσίε εντοπισμού θέσης που παρέχουν ε, οι δορυφορικέ υπηρεσίες. Είδαμε και τα ζητήματα προστασίας δεδομένων, προστασίας ιδιωτικής σφαίρας. Θα σας πω τώρα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Ζήτησε το Συμβούλιο χρησιμοποιήσουμε το 112 ε, να είναι η βάση για όλη τη συζήτηση. Μειώνεται το πεδίο εφαρμογή μόνο στο βασιζόμενο στο 112 ή e call, ε, την, την κλίση αυτή, Θέλουμε επίσης να είναι μόνιμα ενσωματωμένο αυτό το σύστημα στα οχήματα. Εκφράσαμε επίσης την προθυμία μα να δεχθούμε και πρόσθετου ορισμούς που σχετίζονται με υπηρεσίε από τρίτου, με κατάλληλη όμω επεξήγηση της διαφορές μεταξύ του υποχρεωτικού και των εθελοντικών προαιρετικών λύσεων ή η πιθανή συνύπαρξη αυτών επέκταση του πεδίου σε εξαρτήματα ή σε ξεχωριστέ τεχνικές μονάδες. Ό,τι φαίνεται θα είμαστε σε θέση να καταλήξουμε σε μια κοινή προσέγγιση σε ό,τι αφορά τη συμβατότητα με τις υπηρεσίε εντοπισμού θέσης που παρέχουν ε, τα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης. Επίσης, ε, είχαμε δύο συναντήσεις τεχνικής φύσεως μέχρι στιγμής, 16 και 22 Οκτωβρίου συγκεκριμένα. Σε αυτές τις δύο συναντήσεις όλα τα θέματα που δεν θεωρήθηκαν πολιτικές προτεραιότητες και συμπεριλαμβάνονται στο τετράστιλο έγγραφο ε, συζητήθηκαν και δύο ε, οι ορισμοί, το παράρτημα, οι τεχνικές απαιτήσει και τα πρότυπα, τα ε, εναπομένουσες εκλογικές γεύσεις και τα υπόλοιπα. Δεν έχουμε λάβει βέβαια την τελικό feedback το Συμβούλιο για τα τεχνικά ζητήματα. Το Συμβούλιο όμως ήδη έδειξε ότι δέκτυα θετικά στα περισσότερα από τα ζητήματα που εξετάσαμε. Χθες είχαμε μια επίσημη συνεδρία των συντονιστών, των σκιωδών, συγγνώμη, όπου εκεί συζητήσαμε και συμφωνήσαμε την διαπραγματευτική μας θέση για το δεύτερο ανεπίσημο τριμερή διάλογο, ο οποίος ε, θα διεξαχθεί 11 Νοεμβρίου, την επόμενη Τρίτη δηλαδή. Και θα συζητηθούν τα εξή. Πρόσβαση σε ανεξάρτητους παρόχους ε, και πλατφόρμες, περιοδικές τεχνικές επιθεωρήσεις, ε, αναβαθμίσεις υποδομών, και σχετική υποβολή αναφορών, επέκταση σε άλλες κατηγορίες οχημάτων και τελευταίο και σημαντικό βέβαια εξίσου θέμα, ημερομηνία έναρξη ισχύω. Θα επανέλθουμε ε, και στο θέμα της προστασίας δεδομένων και στην ιδιωτική σφαίρα άρθρο 6. Επανειλημμένως έχουμε πει στο Συμβούλιο ότι το άρθρο 6 είναι μια από τις βασικές μας προτεραιότητες στο φάκελο αυτό και ελπίζω γι' αυτό το λόγο το Συμβούλιο να δεχθεί όλες τις τροπολογίες μας που τις έχει η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ να του πρώτου μας διαλόγου. Λίγα είναι τα εκρεμή ζητήματα. Χθες τα συζητήσαμε όλα με τους Σκιώδης και συμφωνήσαμε ότι η διαπραγματευτική εντολή θα προτείνει με τη διπλωματική μα εντολή θα προτείνουμε για, για κάποια, ε, θα κάνουμε προτάσει στο Συμβούλιο για τέσσερα άρθρα και για κάποια συντολικέ σκέψει. Θέλω να ευχαριστήσω όλου του συναδέλφου τη διαπραγματευτικής ομάδα ε, του Κοινοβουλίου αλλά και του ομολόγου μα από Συμβούλιο και Επιτροπή. Ήταν πολύ θετικό το κλίμα. Βέβαια, οι διαπραγματεύσει ήταν αρκετά σκληρέ, ήταν όμω και επικοδομητικέ. και νομίζω ότι όλες οι πλευρές ενδιαφέρονται να επιτύχουμε συμφωνία. Επί Ιταλικής Προεδρίας ελπίζουμε. Ευχαριστώ. Σχόλια παρακαλώ ε, σε σχέση με τα, από τα μέλη μάλλον της ομάδας το ECOM. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω και τους ε, δύο εισηγητές και τη γραμματεία που ασχολήθηκαν με ορισμένα ζητήματα τεχνικής υφής σε λεπτομέρεια και συνεργάστηκαν γιατί προσπαθούμε να συνεργαστούμε και με άλλες επιτροπές γιατί αν είναι πολύ καλή η φήμη μας ως Επιτροπή Συνεργασίας σε αυτό το στάδιο εργασιών, αυτό θα είναι ευεργετικό για εμάς τα επόμενα χρόνια. Δεν θα συμφωνήσουμε στα πάντα. Αν συμφωνούσαμε στα πάντα δεν θα ήμασταν πολιτικοί. Μπορούμε όμως να συνεργαστούμε και να ακούσουμε και τις ανησυχίες από άλλες επιτροπές έτσι ώστε να ασχοληθούμε με αυτά τα ζητήματα εκεί όπου μπορούμε. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία για την φήμη της Επιτροπής. Μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε προσχέδιο γνωμοδότησης για την πολιτική ανταγωνισμού Πρόκειται για έκθεση πρωτοβουλίας, γνωμοδότηση για, το, ε, για την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ε, Επιτροπή Ανταγωνισμού, έκθεση ε, οίκων, καταρχήν. Αυτή είναι η κύρια Επιτροπή. Και ο κύριος Κάλλας... Η κυρία Κάλλας είναι υπεύθυνη και θα της δώσω το λόγο για να μας ε, μιλήσει για το θέμα αυτό, για την έκθεση πρωτοβουλίας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Πιστεύω ότι η ίδια η γνωμοδότηση είναι αρκετά σαφής ως προς το χρονοδιάγραμμα. Είπαμε για να είμαστε έτοιμοι πριν από την Επιτροπή Οίκων, πριν ψηφίσει για την έκθεση η προθεσμία για τις τροπολογίες ε, θα ισχύσει για τις 4 Δεκεμβρίου και στις 22 Ιανουαρίου θα γίνει ψηφοφορία στην Οίκον. Ως προς το περιεχόμενο θεωρώ ότι η πολιτική ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμβαδίζει με οποιαδήποτε νομοθεσία περί εσωτερικής αγοράς, άρα η πολιτική μας αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς που διαδραματίζει κύριο ρόλο για την ε, ίδια τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Γι' αυτό υπογράμμισα στη γνωμοδότηση στη, τη σημασία της ε, καλής συνεργασίας μεταξύ της ε, Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού και της Επιτροπής ε, ΙΜΚΟ. Η ετήσια έκθεση της Επιτροπής σχετίζεται με πολλά ζητήματα. Θα επιθυμούσα να μιλήσω για πολλές από αυτές τις πτυχές, αλλά θεωρώ ότι πρόκειται για αρμοδιότητες της Επιτροπής Οίκων, όπως οι κρατικές επιδοτήσεις και η φορολόγηση που είναι αρμοδιότητες της Οίκων. Γι' αυτό θα, ήθελα να σταθούμε στις δικές μας αρμοδιότητες, αρμοδιότητες της ΙΜΚΟ ως προς τις τροπολογίες. Τόνισα τον ψηφιακό τομέα γιατί θεωρώ ότι μία πιο στεναρή πολιτική ανταγωνισμού χρειάζεται για την ολοκλήρωση της ενιαίας ε, αγοράς. Ως προς το, την Google θα ήθελα να πω ότι υπήρξε μία δήλωση από την Google που ανέλαβε δεσμεύσεις αλλά η Επιτροπή δεν δέχτηκε αυτές τις δεσμεύσεις από την Google Γι' αυτό θα ε, ήθελα να υποβάλω τροπολογία για να διορθώσω τα δεδομένα. Στόχος μας δεν είναι πολιτικός ε, καθαρά σε σχέση με την πάγια νομολογία. Θα θέλαμε όμως η Επιτροπή να διασφαλίσει ώστε οποιαδήποτε απόφαση να επιλύσει το πρόβλημα σε σχέση με την καινοτομία των ΜΜΕ. Γι' αυτό θα ήθελα να ακούσω τα δικά σας σχόλια και απόψεις και ελπίζω να έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Αντρέας. Αντρέας, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα ως και ο από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να ευχαριστήσω τη συνάδελφο Κάλλας. Ε, είναι πολύ καλή ε, η σύνοψη που έκανε ε, για τα θέματα που ενδιαφέρουν την Επιτροπή μας ως προς τον ανταγωνισμό. Υπάρχουν όμως μερικά σημεία που χρειάζονται βελτίωση, ίσως με τροπολογίες, ίσως με συζητήσεις. Το κείμενο ε, το δικό μας είναι γνωμοδότηση, επί της ουσίας είναι αρμόδια οικονομική επιτροπή, θα πρέπει λίγο να το αλλάξουμε. Ε, ο κατακαιρματισμός στην ψηφιακή εσωτερική αγορά είναι κάτι που το θεωρώ σημαντικό. Ταυτόχρονα όμως τίθεται για μένα το εξής ερώτημα. Η ουδετερότητα του δικτύου είναι άραγε ένα θέμα ελέγχου του ανταγωνισμού ή μήπως κυρίως ε, νομοθετικά έχει σημασία. Καλά, μπορούμε να το συζητήσουμε. Στο τέλος να βρούμε τη σωστή διατύπωση. Ε, ίσως και να τσακωθούμε γι' αυτό. Στο σημείο 2 είναι πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρεται για τις μηχανές αναζήτησης. Εγώ προσωπικά είμαι κατά του να κατονομάζονται εταιρείε. Όταν μιλάμε για μηχανές αναζήτησης ξέρουμε τι εννοούμε και ποια δικαστική υπόθεση. Ε, και ποια διαδικασία. Η κυρία Κάλλας το είπε και το διόρθωσε, ε, δεν ήταν σωστό αυτό που γινόταν μέχρι τώρα, γιατί δεν υπήρχε συμφωνία μεταξύ ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Google. Δεν έχει διακανονιστεί αυτή η υπόθεση. Και επίσης νομίζω είναι σημαντικό να έχουμε ως αφορμή και ευκαιρία αυτή τη δικαστική υπόθεση για να δούμε ε, πόσο έχει μετακινηθεί το δίκαιο ανταγωνισμό από την αρχική του ε, πορεία. Ε, βάσει του άρθρου 9, όλο και περισσότερες διαδικασίες καταλήγουν σε διακανονισμό και φιλικό και όλο και λιγότερα μπαίνουν στο άρθρο 6 που συγκρούονται, οπότε αυτοί που φοβούνται αρνητικές ε, αποφάσεις του δικαστηρίου και οι καταναλωτές ε, μπορούν να κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος ε, και μπορούν να προσφύγουν στο δικαστήριο. Σε περίπτωση διακανονισμού όμως καταργείται αυτή η δυνατότητα και για τους καταναλωτές, οπότε θα πρέπει να δούμε μακροπρόθεσμα ποια πορεία πρέπει να ακολουθήσει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού. Και ο Γενικός Εισαγγελέας στο ΔΕΚ που είναι Ολλανδός, είπε ότι ε, παρακολουθεί αυτή την εξέλιξη επίσης με μεγάλη ανησυχία. Όλα αυτά μπορεί να σας φαίνονται πολύ τεχνικά, αλλά αξίζει να τα δούμε σε μεγαλύτερο βάθος ως Επιτροπή ΙΜΚΟ. Η οδηγία τώρα για την εφαρμογή των ε, ε, αξιώσεων για αποζημίωση, ιδιαίτερα σε συλλογική δράση, και συλλογικές ζημίες ε, δεν έχει καταλήξει. Αυτή τη βδομάδα πρόκειται να εξεταστεί. Ελπίζω τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν όλα αυτά όσο γίνεται πιο γρήγορα και πιο ενιαία. Και σε ό,τι αφορά τώρα τις δημόσιες συμβάσεις, θα ήθελα να ασχοληθούμε αργότερα με αυτό το θέμα. Ίσως κάνω και τροπολογίες προσωπικά. Και μπορεί να περιμένει σύντομα τις τροπολογίες μου η συγκεκριά. Sorry, Lucy Anderson. Anderson. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια Κάλλας, ιδιαίτερα για την εργασία της και διότι πολύ γρήγορα συνέταξε αυτή τη γνωμοδότηση, κάτι που μας βοήθησε ιδιαίτερα. Σε σχέση με τα ε, ιδιαίτερα σημεία που θα ήθελε να θίξει η σοσιαλιστική ομάδα, θα πρέπει να σας πω ότι η προστασία του καταναλωτή είναι ύψης της σημασίας και πρέπει να ενισχυθεί σε σχέση με αυτή τη γνωμοδότηση. Επίσης, τασόμαστε υπέρ της προώθησης της ενιαίας ψηφιακής αγοράς και του ανοίγματο αυτού του τομέα, αλλά νομίζω ότι χρειάζονται σαφείς κανόνες ανταγωνισμού και ίσως υπάρχει έλλειψη στοιχείων ως προς την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, προσφυγή στη δικαιοσύνη που είναι πολύ μεγάλη σημασία και εδώ θεωρώ ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε τα δικαιώματα του καταναλωτή. Σε σχέση με τις δημόσιες προμήθειες θα θέλαμε να υπάρχει πρόσβαση στην εξωτερική αγορά ως προς τις δημόσιες προμήθειες. Καταλαβαίνουμε τη συλλογιστική αυτού του υπερβολικού συγκεντρωτισμού στις αγορές του δημόσιου τομέα, αλλά πιστεύω ότι οι μεγάλοι φορείς ε, τα νοσοκομεία και τα σχολεία θα πρέπει να μπορούν να προσφεύγουν άμεσα στην εξωτερική αγορά για να μειώσουν το κόστος. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι άμεσα ε, ε, θέμα της εντολής μας, αλλά θέματα απασχόλησης καθώς και κοινωνικά ζητήματα άπτονται της ε, πολιτικής ανταγωνισμού. Επίσης, οι κρατικές ενισχύσεις είναι κάτι το ξεχωριστό, αλλά δεν μπορούμε να το διαχωρίσουμε, ιδιαίτερα στο τομέα των μεταφορών. Εδώ χρειάζονται κατευθυντήριες γραμμές. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να διαχωρίσουμε από την πολιτική ανταγωνισμού. Ελπίζω να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε τις επερχόμενες εβδομάδες. Ευχαριστώ. Ε, Ο Ντένις Γιόγκ αποσιάζει. Ο Μάρκος επίσης. Η Μαρία Γκραπίνη, θα ήθελα και εγώ να πω ότι εκτιμώ την εργασία της κυρίας Κάλλας. Συμφωνώ με τα σημεία 4 και 5 και συμφωνώ με την προλαλή σε σχέση με το σημείο 6. Για τις ΜΜΕ είναι δύσκολο να έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη ε, λόγω κόστους και τεκμηρίωσης. Και νομίζω ότι πολύ λίγες ΜΜΕ έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Ιδιαίτερα σε περίπτωση του ανταγωνισμού δεν μπορούν να αντιδράσουν και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να απλουστεύσουμε την ε, πρόσβαση στην τεκμηρίωση και να ασχοληθούμε και με το θέμα του κόστους. Στα σημεία 4 και 5 έχει σημασία η διατύπωση. Γιατί νομίζω ότι παραμένει το πρόβλημα των δημόσιων αγορών. Οι δημόσιες προμήθειες, όπως είπε και η προλαλή σας, αφορούν μεγάλες ποσότητες, δηλαδή μεγάλες συμβάσεις όπου οι ΜΜΕ ε, δεν έχουν πρόσβαση. Όταν ήμουν υπουργό στη Ρουμανία προσπάθησα να αντιμετωπίσω αυτό το θέμα γιατί προσπαθήσαμε να κάνουμε μια περιφερειακή κατανομή αγορών στον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης έτσι ώστε οι ΜΜΕ να έχουν πρόσβαση γιατί ο κύκλος εργασιών έτσι είναι μικρότερος όταν γίνεται αυτή η κατανομή. Γιατί πιστεύω ότι δεν έχει σημασία μόνο ο ορισμός ή οι ορισμοί, αλλά το πώς γίνονται οι δημόσιες ε, προμήθειες. Γιατί εάν θεωρώ ότι ότι, ότι υπάρχουν ε, ή έχουμε να κάνουμε με αστρονομικά ποσά, δεν ε, προσπαθούν, δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση οι ΜΜΕ. Τουλάχιστον αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε στη Ρουμανία, να κατακαιρματίσουμε τις μεγάλες συμβάσεις σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ιδιαίτερα για τα σχολεία και τα νοσοκομεία. Άρα τα σημεία 4 και 5 δεν αρκούν. Θα πρέπει να υπάρχει εποπτεία των δημοσίων προμηθειών. Στη Ρουμανία διαπιστώσαμε ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις ε, τι έκαναν, αναλάμβαναν ένα έργο και μετά ε, προέβαιναν σε υπεργολαβίες. Και υπήρχαν μεγάλα προβλήματα. Άρα ο συγκεντρωτισμός που βοηθάει δεν έχει νόημα για τις δημόσιες προμήθειες. Υπάρχει όμως ε, προγραμματισμός και αυτό που έχει σημασία είναι ποιος μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον στους ε, διαγωνισμούς. Γι' αυτό αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ρύθμιση του πλαισίου και νομίζω ότι με αυτή την έκθεση θα μπορούσαμε να αλλάξουμε κάτι γιατί οι δημόσιες προμήθειες είναι μία μακροχρόνια ιστορία. Δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τις ΜΜΕ παρά με μία νέα πλαισίωση των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ, λέει ο μου φαίνεται καλή προσέγγιση σε ό,τι αφορά την ενημέρωση για τις αρχές, όχι μόνο τις αρχές ανταγωνισμού, αλλά για παράδειγμα και τις αρχές προστασίας δεδομένων. Θα πρέπει να είναι διαθέσιμες και διαφανείς οι πληροφορίες αυτές, ιδίως σε ό,τι αφορά την, ε, τον τρόπο επεξεργασίας των πληροφοριών. Δεν είναι ξεκάθαρο μέχρι στιγμής τι ακριβώς γίνεται και συχνά οι αρχές δεν είναι καν σε θέση να ελέγξουν εάν οι υπηρεσίες αυτές ενεργούν με γνώμονα τους ε, κανόνες της ε, εσωτερικής αγοράς. Και αυτό το δεύτερο σημείο μου, γιατί νομίζω ότι καλό θα ήταν, δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη όλοι, στην απόφαση του Μαΐου του τρέχοντος για τις μηχανές αναζήτησης και την υποχρέωση να σέβονται τους κανόνες περί προστασίας δεδομένων όπως είναι η του 95 Καθίσταται σαφέ λοιπόν σε αυτή την απόφαση ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνε ισχύουν για τι υπηρεσίε αυτέ, ακόμη και αν προέρχονται εκτό ευρωπαϊκών αγορών. Δηλαδή μπορεί η έδρα τη επιχείρηση να είναι εκτό Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά παρόλα αυτά οι ευρωπαϊκοί κανόνε ισχύουν. Και γι' αυτό πρέπει και εδώ να αναφερθεί ότι, γίνεται, ε, ότι είναι ανάγκη να γίνονται σεβαστά τα ευρωπαϊκά πρότυπα και οι κανόνες, όπως ε, οι κανόνες περί προστασίας δεδομένων. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, Εύελιν Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και την κυρία Κάλλας. Είναι πραγματικά πολύ καλό το κείμενο που μας έδωσε. Και πιστεύω ότι βάσει αυτού μπορούμε να εργαστούμε πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν δύο σημεία που θέλω να αναφέρω στόσο και επιβεβαιώνω και τονίζω αυτά που είπε η Λούση Άντερσον, συνάδελφος και σκιώτης ηγήτρια της ομάδας μου, ότι θα πρέπει λίγο περισσότερο να συμπεριλάβουμε ε, τον τομέα της προστασίας καταναλωτού ε, και το σημείο 4, γιατί εκεί στις δημόσιες συμβάσεις ε, το θέμα δεν είναι μόνο η καλύτερη σχέση τιμής ε, και προσφοράς. Δεν θέλουμε μόνο τη πιο φθηνή προσφορά, το μειοδότη ας πούμε, αλλά και την καλύτερη που λαμβάνεται υπόψη η προστασία των καταναλωτών, του περιβάλλοντος ή και κάποια άλλα δικαιώματα. Είναι και αυτά στοιχεία που πρέπει να συνυπολογίζονται και οπωσδήποτε να τα ενισχύσουμε κάπως. Ζήτησα όμως το λόγο προηγουμένως και για κάτι που είπε ο συνάδελφος Ανδρέας Φαπ, ο οποίος δυστυχώς αποχώρησε, αλλά θα το πούν οι βοηθοί του. Είναι ένα σημείο στο οποίο διαφωνώ μαζί του, ότι η ουδετερότητα ε, του δικτύου ε, ε, λέει, δεν έχει να κάνει με το διαδίκτυο, δεν έχει να κάνει με τον ανταγωνισμό, μα η ουδετερότητα του δικτύου είναι ακριβώς προϋπόθεση για να έχουμε δικαιοσύνη και στον ανταγωνισμό. Και πολύ σωστά η κυρία Κάλλας ε, μιλάει για αυτό το θέμα και με τέτοια σαφήνεια το έχει γράψει κιόλας. Και γι' αυτό δεν θα το θεωρούσα ε, σκόπιμο ούτε καλό να το βγάλουμε ή να το σχετικοποιήσουμε ή να το αποδυναμώσουμε ανάλογα με τις τροπολογίες του κυρίου Σφάπ. Κατά τα άλλα πιστεύω ότι ως ομάδα μπορούμε να ασχοληθούμε και με τον ανταγωνισμό και την προστασία των καταναλωτών οπωσδήποτε και να ενισχύσουμε στο κείμενο το το περισσότερο. Ευχαριστώ. Any other speakers? Άλλοι ομιλητές. which case... Όχι. Θα ήθελα και εγώ να υποβάλω μερικά σχόλια στην ετήσια έκθεση για τον ανταγωνισμό θα έχουμε πολλές γνωμοδοτήσεις από πληθώρα επίτροπων και η εισηγήτρια μας είπε ότι εμείς θα πρέπει να παραμείνουμε στις δικές μας αρμοδιότητες. Αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί αν αρχίσουμε να σχολιάζουμε για ζητήματα που σχετίζονται με τις κοινωνικές υποθέσεις ή την αποσχόληση τότε υποβάζουμε το ρόλο μας. Αν θέλετε να υποβάλλετε σχόλια για αυτά τα ζητήματα, να το κάνετε, αλλά στις αρμόδιες επιτροπές. Η δική μας έκθεση θα πρέπει ε, να λάβει υπόψη, να ασχολείται μόνο με θέματα δικών μας αρμοδιοτήτων. Ως προς το ψηφιακό τομέα, θα πρέπει να μιλήσουμε για τον διαχωρισμό ε, φορέων, unbundling, και να δούμε και τα ε, ωφέλη ομότιμων, ομότιμων αρχών εναντί των καταναλωτών για να υπάρχει ίση ε, πρόσβαση στην αγορά τη στιγμή που πρόκειται για κανόνες μεταξύ ομοτήμων. Υπάρχουν αρκετοί τομείς όπου θα μπορούσε το Κοινοβούλιο να νομοθετήσει στον ε, ψηφιακό τομέα όπου να υπάρχει λιγότερος ανταγωνισμός και όχι περισσότερος. Και εδώ λαμβάνω υπόψη τα συστήματα πληρωμών τα οποία θα μπορούσαν να απορροφήσουν τα μονοπόλια και να ενθαρρύνουν τον ανταγωνισμό. Και εδώ μιλώ και για τις μεθόδους ε, πληρωμών στον χρηματοοικονομικό τομέα. Συμφωνώ με τους προηγούμενους ομιλητές όταν μίλησαν για ευεργετικά σχήματα σε σχέση με το σημείο 2. Δεν θα πρέπει να προδικάσουμε τις αποφάσεις ε, του τρόπου ανταγωνισμού γιατί θα πρέπει να πρόκειται ε, για ανεξάρτητες ε, αποφάσεις χωρίς πολιτική χρειά. Ως προς τα άρθρα 4 και 5 για τις δημόσιες προμήθειες, Πιστεύω ότι οι νομοθετικές αλλαγές ε, έγιναν κατά την τελευταία θητεία και υπήρχε μεγάλη πολιτική συμφωνία από όλες τις πολιτικές ομάδες και κόμματα. Γι' αυτό θα πρέπει οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να συμμετάσχουν και στις μεγάλες και στις μικρές συμβάσεις και να μην ε, υπάρχουν μονοπόλια. Να ενθαρρύνουμε την καινοτομία. Αλλά ας μην επαναλάβουμε την εργασία η οποία έχει λήξει. Θα μπορούσαμε από την Επιτροπή να μας δώσει διασαφήσεις για το πώς λειτουργεί έμπρακτα η νομοθεσία για τις δημόσιες προμήθειες ιδιαίτερα για τις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις που θεωρούν ότι θα μπορούσαν να αναλάβουν μια σύμβαση ή θα μπορούσαν να προβάλλουν περισσότερη καινοτομία. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να έχουμε έναν πιο εύρωστο δημόσιο τομέα. Θα πρέπει να ζητήσουμε διευκρινήσεις από την Επιτροπή εμείς είμαστε η Επιτροπή που ε, θεωρεί ότι στο εμπροστοφυλακή είναι οι καταναλωτές, καταπολεμούμε τα καρτέλ, λαμβάνουμε υπόψη τις ε, ζημίες που υφίστανται οι καταναλωτές και ε, έχουμε υποβάλει και τροπολογίες επί του θέματος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ε, γιατί παρά το, το γεγονό ότι η έκθεση αυτή ήταν περιορισμένη και από πλευράς μεγέθους τα καταφέρατε πολύ καλά. Θέλει κάτι να πει η συγγήτρια. Εν... Σύντομο σχόλιο αν με επιτρέπετε. Προσβλέπω στις τροπολογίες σας, τα σχόλιά σας και τώρα ε, να αναφέρω και δύο-τρία πράγματα. Σε ό,τι αφορά τι κρατικέ ενισχύσει, για παράδειγμα, συμφωνώ. Πρόκειται για μια βασική πολιτική στον τομέα του ανταγωνισμού. Αλλά είναι και αρμοδιότητα τη ΕΚΟΝ και εξού το άφησα εκτό. Οι κρατικέ ενισχύσει στον τομέα των μεταφορών είναι ένα άλλο παράδειγμα. Θα το ε, εξετάσει αυτό η Επιτροπή Αναφορών σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και τα σχετικά. Είναι αρμόδια της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ που θα ασχοληθεί επομένως και με αυτήν την πτυχή, έξω και δεν το αναφέρω εδώ. Τουλάχιστον όχι τόσο διεξοδικά. Συμφωνώ ότι ίσως καλό θα ήταν να μην κατονομάζονται επιχειρήσεις, να παραμείνουμε σε γενικόλογες διατυπώσεις. Ε, άρα θα προβώ σε σχετική τροπολογία, τροποποίηση. Σε ό,τι αφορά τις δημόσιες συμβάσει, Συμφωνώ ότι ναι μεν τέθηκε πρόσφατα σε ισχύ, άρα πρέπει να αφήσουμε λίγο χρόνο για να γίνουν κατανοητοί οι κανόνες και να εφαρμοστούν. Αλλά πρέπει και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να καταλάβουμε ότι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν. Αυτά λοιπόν. Ευχαριστώ όλες και όλους για τα σχόλια. Πρόεδρος. Εγώ ευχαριστώ. Να σας υπενθυμίσω την προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών 4 Δεκεμβρίου. 21 και 22 Ιανουαρίου ψηφίζουμε εδώ στην Επιτροπή μας. Ίσως ζητήσω να λάβει τις σχετικές διευκρινήσεις η συγκήτρια για το τι θα συμβεί αν υποβληθούν από την Επιτροπή μας τροπολογίες που είναι καθαρά εκτός του πεδίου αρμοδιότητάς μας. Μπορεί να θεωρηθούν μη παραδεκτές ή όχι. Ε, αν υπάρχουν θέματα, μιλήστε παρακαλώ με τους συναδέλφους σας από τις άλλες επιτροπές που έχουν και αυτές να συντάξουν εκθέσεις για το θέμα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπω ότι προχωράμε πιο γρήγορα από ό,τι προβλέπετε στην ημερήσια διάταξη και αυτό είναι πολύ καλό. Αν συμφωνείτε, όσοι συναδελφοί είστε παρόντες, έχουμε μια παρουσίαση τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η οποία θα μας μιλήσει για το κόστος και την χρησιμότητα του Container Status Message αυτού του συστήματος. is the nice man who's taking the pictures. Να και ένας καλός κυριούλης που με παίρνει φωτογραφίες. I'm just checking because the EPP ήθελα να ελέγξω γιατί δεν βλέπω σκιώδη από το ΕΛΚΑ. Από τις άλλες ομάδες όμως βλέπω, άρα δεν ξέρω, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Μάλιστα. Επομένως, να καλωσορίσω στην Επιτροπή μας του Μάρκοτ Χόφμαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα μας παρουσιάσει αυτή την πρόταση. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Επαναλαμβάνω, ουσιαστικά είναι μία μελέτη για τα συμπεράσματα που ε, προέκυψαν από τη μελέτη των στοιχείων του κόστους και της χρησιμότητας της υπηρεσίας ε, τα μηνύματα κατάστασης εμπορευματοκιβωτίων. Container status messages. Υπάρχουν μηνύματα όταν κάτι στην Ευρώπη. Το θέμα είναι κατά πόσο θα πρέπει να έχουμε μηνύματα και κατά την εξαγωγή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μας επιτρέπετε να γνωμοδοτήσουμε για αυτό το θέμα, να συστηθώ σύντομα, γιατί για πρώτη φορά έρχομαι στην Επιτροπή σας, Μαργαρέτε Χόφμαν λέγομαι, όπως σωστά είπατε, και είμαι Διευθύντρια στο Τμήμα Πολιτικής για την καταπολέμηση ε, της απάτης στην ε, Όλαφ. Λάθος μικρόφωνο είχα ανάψει, ζητώ συγγνώμη. Μάλιστα. Έλεγα λοιπόν να συστηθώ σύντομα, Μαργαρέτε Χόφμαν λέγομαι και είμαι Διευθύντρια στις πολιτικές Όλαφ, που είναι το γραφείο για την καταπολέμηση της απάτης και παρακολουθούμε τη μεταρρύθμιση του κανονισμού 515 του 97 και είμαστε αρμόδια. Έχουμε με τους συναδέλφους προετοιμάσει μια μικρή παρουσίαση PowerPoint και θα τα παρουσιάσει ε, ο παρακαθήμενος συνάδελφος. Να τα πω στα αγγλικά πρώτα, κάποια εισαγωγικά σχόλια. Ε, με ιδιαίτερη χαρά ερχόμαστε να μιλήσουμε στην Επιτροπή σας σήμερα για αυτό το ειδικό θέμα, ε, για την εξαγωγή στο Container Status Messages. Έχουμε πάντα μεγάλη υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, για την προστασία των χρημάτων των φορολογουμένων, είτε πρόκειται για τα έσοδα είτε για τις ε, δαπάνες. Και αυτό είναι κάτι που ενδιαφέρει και την Όλαφ και το Κοινοβούλιο. Έχουμε ε, γίνει πολλές πρόοδοι στην εσωτερική αγορά και πολλοί, πολλές επιχειρήσεις δηλαδή έχουν σχεδόν απρόσκοπτη διασυνοριακή δράση και θα πρέπει να υπάρχουν τα απαραίτητα εργαλεία ε, διασυνοριακά για να διώκεται η απάτη με τρόπο αποτελεσματικό. Και γι' αυτό το λόγο πέρυσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως όλοι γνωρίζετε ε, πρότεινε ε, μια σειρά βελτιώσεων στο βασικό ε, κανονισμό 51597 που έχει διάρκεια ζωής άνω της 15 ετίας και καλό θα είναι να εξυγχρονίζεται και να συμβαδίζει με τις σύγχρονες τεχνολογίες για να απαντά ε, στα νέα σχήματα απάτης που εμφανίζονται. Ε, τα παραθυράκια και οι αδυναμίες δημιουργούνται από την έλλειψη πληροφοριών και αυτά οι απαταιώνες τα εκμεταλλεύονται με ε, απώλεια εισοδήματος και για τα κράτη-μέλη και για τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Για να κλείσουμε λοιπόν αυτά τα παραθυράκια τι πρέπει να κάνουμε. Και θέλω να τονίσω και έχει σημασία για μας οι τροποποιήσεις που προτείνουμε δεν έχουν σχεδιαστεί μόνο για να βοηθήσουν την Όλαφ ή την Κομισιόν για να καταπολεμήσει την τελωνιακή απάτη. Ε, είναι πολύ σημαντικό, ακόμα και σημαντικότερο για να θωρακίζονται τα κράτη-μέλη για να προστατεύουν τα φορολογικά έσοδα. Η καταπολέμηση λοιπόν των τελωνιακών απατών στους δασμούς είναι συναρμοδιότητα και καλό θα είναι να έχουμε κοινή προσπάθεια για να το αντιμετωπίσουμε. Είμαστε πολύ ευγνώμονε για την υποστήριξη που μα έχετε δώσει εσεί και τα κράτη-μέλη σε πολλέ από τι τροποποίησει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα επίση να σα ευχαριστήσω και τους ε, εισηγητές του Κοινοβουλίου και το προηγούμενο και τον ΙΝ για την ταχύτητα με την οποία αντέδρασε. Είμαστε αρκετά ε, προχωρημένοι και προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε την προσπάθεια αυτή πριν τα τέλη του έτους. Σήμερα θέλουμε να σας δώσουμε περισσότερες διευκρινήσεις για ε, την διάδοση πληροφοριών και διαβίβαση για τις εξαγωγές. Ξέρω ότι ενδιαφέρει πολλούς από εσά και σε πρώτη ανάγνωση το Κοινοβούλιο δεν συμπεριέλαβε, όπως πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, της ΕΣΜ ε, ε, των εξαγωγών. Γι' αυτό Χαιρόμαστε που έχουμε την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε εδώ σήμερα τις απόψεις μας. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάφερε να εξηγήσει στα κράτη-μέλη, στο Συμβούλιο, την ακριβή φύση αυτού του ε, θέματος που προτείνουμε. Προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι αυτό που προτείνουμε δεν σημαίνει επιπλέον άχρηστο γραφειοκρατικό άχθος για τον κλάδο, για τις επιχειρήσεις, αλλά είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο για την καταπολέμηση ε, της απάτης. Ε, επί της ουσίας τι προτείνουμε. Υπάρχουν ήδη οι ε, ηλεκτρονικές προφορίες από τις ναυτιλιακές εταιρείες και που θα πρέπει να στέλνονται ε, στην ε, Όλαφ. Βεβαίως πάντα με ό,τι ισχύει για την εμπιστευτικότητα και το απόρριτο. Χαίρομαι που το Συμβούλιο καταρχήν συμφώνησε με τα όσα εμείς προτείνουμε και η θέση που έλαβε υποστηρίζει το βασικό κορμό της πρώτας Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα δεδομένα και τα CSM των εξαγωγών. Επίσης είμαστε σε επαφή και με τις ναυτιλιακές εταιρείες για να τους εξηγήσουμε καλύτερα τι εννοούμε. Κατανοούμε ότι η αρχή λοιπόν δεν είναι κάτι το οποίο αφισβητεί ούτε ο κλάδος ο ίδιος ο ναυτιλιακός. Βεβαίως Παραμένουν κάποιες ανησυχίες και το παραδέχομαι. Θα σας εξηγήσει ο κύριος Ράις, ο, ο συνάδελφος, στη συνέχεια. Θα ήθελα να υπογραμμίσω και πάλι ότι η απάτη δεν συμβαίνει μόνο στις εισαγωγές, όπου οι δασμοί και ε, φόροι οφείλονται. Εξίσου ε, επιρρεπές ε, σε απάτη είναι και το σύστημα εξαγωγών μας. Θα σας εξηγήσει λοιπόν ο κύριος Ράις πώς τα δεδομένα των εξαγωγών και τα CSM μπορούν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της απάτης στα τελωνία. Είναι και το απογραμμίζω ένα νέο βήμα στην καταπολέμηση της απάτης, αλλά ε, είναι οπωσδήποτε απαραίτητο και απολύτω και αν συμφωνείτε θα παρακαλέσω τον κύριο Ράις να εξηγήσει αυτά τα θέματα. Είναι μικρή η παρουσίαση σύντομη, 9-10 διαφάνειες, αλλά ε, θα σας βοηθήσει πραγματικά. Ευχαριστώ. So thank you very much Just for me the... quickly, these oh. slides are available through... Υπάρχουν διαθέσιμες οι διαφάνειες αυτές και μάλιστα και online. On your devices. On the, on the e-meeting. No? Yes. So thank you very much for giving me the... Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Θα έρθω κατευθείαν στην ουσία. Αυτά τα μηνύματα λοιπόν συνδυαζόμενα με δεδομένα έξοδος θα μπορούσαν να να βοηθήσουν να καταλάβουμε μήπως υπάρχουν κάποιες εισαγωγές που είναι παράνομες. Είναι χρήσιμο λοιπόν για στοχευμένους ελέγχους και για την επαλήθευση προορισμού κάποιων ευαίσθητων εξαγωγών και έχω για κάποια παραδείγματα. Έχουμε συλλέξει εμπειρία στον τομέα αυτό μέσω του Contrafic, είναι ένα project που στόχο έχει τη συλλογή αυτών των μηνυμάτων ε, και υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη που ήδη συμμετέχουν. Στο πλαίσιο αυτού του project ε, στείλαμε ένα ερωτηματολόγιο στα κράτη-μέλη, συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του 2013, συμμετείχαν 280 ε, τελωνία και το 20% περίπου δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν και για ελέγχους εξαγωγών το σύστημα. 57 τελωνιακοί 18, από 18 κράτη-μέλη έχουν λοιπόν ήδη αρχίσει να χρησιμοποιούν πιλωτικά. Και από τους 54 χρήστες, οι 43 δήλωσαν ότι οι πληροφορίες που έλαβαν τους έδωσαν ε, μεγάλη βοήθεια στη δουλειά τους, άρα ήταν σημαντικές. Το 1 πέμπτο επίσης ε, των ε, χρηστών, των ερωτηθέντων ε, χρησιμοποίησαν και για τους για τις εξαγωγές. Υπάρχει λοιπόν σύγκριση των στοιχείων αυτών, είναι ανοιχτή πηγής, Τα στοιχεία παρέγονται εθελοντικά και στο σχέδιο το project συμμετείχαν 12, αλλά το σύστημα και τα αποτελέσματά του δόθηκαν σε όλες τις διοικήσεις, ελληνικές, διοικήσεις των κρατών μελών. Πριν περάσω στα παραδείγματα με αυτά τα CSM, που περιγράφουν την κατάσταση και τις κινήσεις των εμπορευματοκιβωτίων. Δεν είναι ονομαστικά. Μπορεί να περιλαμβάνουν στοιχεία περί άφηξης, εφόρτωσης, εκφόρτωσης και της σχετικής εγκατάστασης. Αν αυτή η εκφόρτωση έγινε από το πλοίο, τι οδηγίες έλαβε το προσωπικό, αν χρειάστηκε να σταλεί για επισκευή το εμπνευματοκιβώτο και το καθεξής. Βλέπετε στην οθόνη σας ένα πολύ συνηθισμένο σενάριο, παραδείγματος χάρη, εξαγωγή τσιγάρων ε, μέσω, ε, με εμπορευματοκιβώτια. Φτάνουν σε μια τρίτη χώρα τα εμπορευματοκιβώτια, και μετά επαναφορτώνονται στα πλοία και επανέρχονται αλλά με αλλαγμένα έγγραφα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτά τα CSM μπορούμε να δούμε ότι τα αγαθά εξακολουθούν να βρίσκονται σε περιματοκιβώτιο όταν ξαναφτάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι καλό εργαλείο λοιπόν για να εντοπίσουμε αυτού του είδους την απάτη. Um, Δεύτερο παράδειγμα. Κάποιες εταιρείες στα κράτη-μέλη ε, έχουν κάποια συστήματα πατών όπου δηλώνουν πραγματικά ανεδαφικά υψηλές τιμές για τις εξαγωγές. Αυτό είναι η βάση για την επιστροφή του καταβληθέντος ΦΠΑ, απάτη δηλαδή. Ε, και με τα CSM ε, μπορούμε να δούμε κατά πόσον ξεφορτώθηκαν ή όχι τα εμπορεύματα και έπειτα να προχωρήσουμε σε περαιτέρω έλεγχος για να δούμε τι συνέβη με αυτά τα εμπορεύματα έφτασαν πράγματι εκεί που έπρεπε και μπορούμε να κάνουμε και άλλες επαληθεύσεις. Αυτό είναι ένα πραγματικό παράδειγμα. Το ανέφερε πρόσφατα ένα κράτος μέλος και μας δείχνει και αυτό πόσο χρήσιμα είναι αυτά τα μηνύματα όχι μόνο για την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και για τις υπηρεσίες των κρατών μελών. Ο κανονισμός 515 είναι ο κανονισμός που έχουμε στη διάθεσή μας ως εργαλείο και η Κομισιόν βέβαια αλλά και τα κράτη-μέλη για να εξασφαλίσουμε τη σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας για τα τελωνία, για τα γεωργικά ζητήματα, αλλά εδώ μιλάμε για τα τελωνιακά θέματα. Και όταν μιλάμε για αγαθά διπλής χρήση και για τα εμπάρκο, είναι πολύ σημαντικό για τα κράτη-μέλη και για το κοινό βέβαια να ξέρουν ότι τα εμπορεύματα που παράγονται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι φτάνουν στο σωστό προορισμό. Με αυτά τα δεδομένα, με αυτά τα μηνύματα μπορούμε να δούμε πού καταλήγει ένα πνευματοκιβώτιο. Um, of course. Βέβαια δεν σημαίνει ότι αυτό παρεμποδίζει το να καταλήξουν σε λάθος μέρος ε, κάποια εμπορευματοκιβώτια. Αν εφαρμοστεί σωστά όμως τελωνιακή νομοθεσία, ε, ανοίγουν μέτρα για άλλες δράσεις, ε, έρευνες, ε, ελέγχους από κράτη-μέλη και σε άλλους τομείς. Τέταρτο παράδειγμα, ίσως μοιάζει κάπως με το πρώτο παράδειγμα που σας ανέφερα. Περί τίνος πρόκειται. Όταν οι Ιταλονικές αρχές, ένα δεδομένο παράδειγμα, σας δίνω, δεν θέλω να κατονομάσω χώρες, ας πούμε, έρχονται ε, τσιγάρα, μάλλον ε, μεταφέρονται στη Μάλτα. Βλέπουν οι Μαλτέζοι και ελληνικές αρχές ότι φτάνουν τα τσιγάρα. Αλλά είναι σε διαμετακόμιση. Μπορεί να μην προορίζονται κατά ανάγκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρούν ότι δεν πρέπει να κατασκευθούν αυτά τα τσιγάρα, είναι εκεί, αλλά από τη συσκευασία τους φαίνεται ότι δεν έχουν ε, την φορολογική σφραγίδα των κρατών μελών, μπορεί να είναι επομένως προϊόν παράνομης πόλης, μπορεί να είναι λαθρέα. Με το CSM, αυτό το μήνυμα, μπορούμε να δούμε. Φτάσανε στην αναφερόμενη τρίτη χώρα που αναφέρονταν ως προορισμό αυτά τα τσιγάρα. Ή μήπως στην ανοιχτή θάλασσα τα ξεφόρτωσαν ή ε, λίγο πριν φτάσει στον ε, λιμένα το, τον ευρωπαϊκό το οποιο μεταφέρει αυτά τα τσιγάρα, έχουν αλλάξει τα έγγραφα και τελικά εισάγονται λαθρέα αυτά τα τσιγάρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν μιλάμε για κόστος, για αυτά τα μηνύματα. Αυτά τα μηνύματα είναι διαθέσιμα στους ε, μεταφορείς. Οι μεγάλοι μεταφορείς τα έχουν αυτά τα CSM. Κάποιοι μπορούν να έχουν πιο πολλά, κάποιοι λιγότερα ε, μηνύματα. Όπως λέμε όμως και στην νομοθετική πρόταση, εμείς εξετάζουμε τα διαθέσιμα δεδομένα μόνο. Δεν ζητούμε ε, από κανένα να δημιουργήσει νέα μηνύματα ή κάτι άλλο που θέλουμε να συλλέξουμε. Βασίσουμε την πρότασή μας στα υφιστάμενα δεδομένα. Έχουμε την εμπειρία μας, αλλά έχουμε ε, αποταθεί και στον κλάδο. Και για το τι γίνεται στις ΗΠΑ. στο 40% γίνεται το λεγόμενο global dump ε, για όλα τα μηνύματα δηλαδή. Στην τέτοια περίπτωση θα είχαμε μηδενική, ε, μηδενικά έξοδα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είχαν τα στοιχεία και η Κομισιόν, η Όλαφ, θα μπορούσε να εξετάσει ποια έχουν σημασία. Η online πρόσβαση επίσης είναι μια λύση Δηλαδή με πρόσβαση online οι υπηρεσίες της Κομισιόν μπορούν να συλλέξουν τα δεδομένα. Και πάλι σχεδόν μηδενικό το κόστος αφού δίνει πρόσβαση οι διάφορε εταιρείε μεταφορών και οι τελωνικέ του υπηρεσίες. Υπάρχει και μια τρίτη επιλογή. Να οριστεί συγκεκριμένα ποιες, ποια μηνύματα, ποιες πληροφορίες θέλουν οι αρχές. Μια επιλεκτική αναφορά. Αυτό έχει το κόστος της βέβαια, ως μέθοδος. Είχαμε κάποιες συζητήσεις με τη βιομηχανία και με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ναυτιλίας. Σε ό,τι αφορά την υποχρέωση υποβολής αυτών των στοιχείων ε, δεν φαίνεται να αμφισβητούν πια. Καταλαβαίνουν την ανάγκη. Κάποια σημεία παραμένουν προβληματικά, θα μπορούσαν να λυθούν στους επικείμενους τριμερείς διαλόγους ή και με κατεξουσιοδότηση πράξης. Πρόκειται για συμβάντα που κινητοποιούν αυτό το μηχανισμό, ενεργοποιούν ε, αυτά τα μηνύματα. Αναφέρονται συγκεκριμένα κάποια συμβάντα στο κανονισμό, αλλά θα πρέπει να δούμε και να συζητήσουμε τα δικαιώματα πρόσβασης, ποιος έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, πότε θα τεθεί σε ίσχυο ο κανονισμός, σημαντικό στοιχείο για τους μεταφορείς, για τον κλάδο, και το λεγόμενο vessel diversions, δηλαδή κάποια πλοία για εξωτερικούς λόγους φτάνουν σε ένα ευρωπαϊκό λιμάνι που δεν ήταν όμως προγραμματισμένο στο φιλοπορία τους. Έκαναν δηλαδή μια παράκαμψη, εκτροπή από το δρομολόγιο. Αυτά τα θέματα όμως μπορούν να λυθούν πιστεύω. Επομένως, νομίζουμε ότι με τις σκέψεις αυτές φαίνεται ξεκάθαρα ότι και αυτά τα CSM εξαγωγών θα συμβάλλουν ε, και θα είναι και μάλιστα αποδοτικές προς το κόστος για την ανείχνευση παραβάσεων της τελωνιακής νομοθεσίας και θα βοηθήσουν και την έρευνα της τελωνιακής απάτης. Εμείς δεν παρεμβαίνουμε ε, στα νομικά, ούτε ε, καθυστερούμε, ούτε δημιουργούμε προβλήματα σε εμπορευματικές μεταφορές. Απλά θέλουμε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα των ελέγχων. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Um, Ευχαριστούμε πολύ τους Χόφμαν και Ράις για τις ε, παρουσιάσεις αυτές. Θα ε, δούμε τους ΙΤΕΣ τους, ε, σε σχέση με την εισήγηση αυτή του Σκιώδης. Ε, Ανδρέας Φαμπ από το ΕΛΚ. Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ Βίκη ο δικός μας σκιώδης ηγητής δυστυχώς κολλείεται και μου ανέθεσε να σας τα πω εγώ. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή περί τίνος πρόκειται. Το θέμα δεν είναι ότι κάνει μια πρόταση όλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην περασμένη θητεία είχε ήδη ψηφίσει την πρόταση αυτή. Και η πρόταση αυτή, όπως την έχουμε ξανά σήμερα στα χέρια μας και μας την παρουσιάζεται, την απορρίψαμε. Και με όλα αυτά που ακούω σήμερα, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και συναρπαστικά και μπορώ να καταλάβω ότι σωστά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θέλει να καταπολεμήσει περισσότερο κάποιο λαθρεμπόριο, αλλά στην τροποποίηση του κανονισμού 515 του 97 αυτό δεν έχει να κάνει την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου τσιγάρων, αλλά πώς βοηθάμε διοικητικά γενικά τα τελωνία για να εφαρμόζουν τις αρχές και τις ρυθμίσεις και τους κανόνες. Και δεν αρκεί απλώς να μιλάμε τώρα για χρησιμότητα, usefulness. Είναι ανάγκη, necessity, αναγκαιότητα. Μέχρι τώρα αυτά δεν τα ακούω εγώ και δεν καταλαβαίνω για ποιον ισχυρό λόγο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποκλίνει ε, από την ε, απόφαση της περασμένης θητείας, που ήταν απόρριψη της πρότασης. Θα ήθελα να πω δύο-τρία ακόμα να προσθέσω. Είναι γεγονός ότι δεν υπάρχει επιπλέον κόστος και επίσης είναι ε, γεγονός ότι δεν βλάπτει το εμπόριο, αλλά εγώ δεν ακούω αρκετά να δικαιολογεί ε, τους άλλους κινδύνους. Βάζουμε πολύ βαθιά το χέρι μας ε, στα ε, δεδομένα του εμπορίου και τους δρόμους του εμπορίου ορισμένων επιχειρήσεων. Υπάρχει θέμα προστασίας των δεδομένων και των εμπορικού απορρίτου. Ε, τι νόημα λοιπόν έχουν οι προτάσεις, τι θα χρησιμεύσουν και ποιες δυνατότητες ε, έχουν, αλλά και ποιους κινδύνους έχουν και ποιες δυσκολίες. Και ως εισηγητή λέει ο κύριος Χέλβικ ότι θα αρχίσει διαπραγματεύσει στο Κοινοβούλιο με το Συμβούλιο μόνο εφόσον ε, αρχίσουν οι συνομιλίες βάσει της ηλυμένης απόφασής μας τη περασμένη θητείας. Θα ελέγξουμε πάρα πολύ αυτά που μας είπατε, αλλά ε, καταρχήν ο εισηγητή μα λέει ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα επί τη ουσία και δεν υπάρχει λόγο να ανατραπεί η λιμένη απόφαση του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Συγγνώμη. Έπρεπε πρώτα να είχα δώσει το λόγο στην κυρία Γιά Κονσάρη. Θέλει όμω να ακούσει πρώτα του Σκιώδη ή να μιλήσει πρώτα εσύ. Ναι, οκ, okay, πρώτα οι σκιώδες. Εντάξει. Uh, Νομίζω ότι η κυρία Κάλλας θα ήθελε να σχολιάσει. Υπάρχουν άλλοι σκιώδεις που θα ήθελα να σχολιάσω Και μετά θα συνοψίσουμε. Η κυρία Κάλλας. Ήθελα να υποβάλω μία ερώτηση. Ελέγχθη ότι τα συστήματα αυτά είναι ε, χρήσιμα για την ανείχνευση περιπτώσεων παραβίασης της κοινωτικής νομοθεσίας. Όμως πώς, ε, πώς έχει κατάσταση σε σχέση με τους γενικούς ε, κανόνες, σε σχέση με τη, την παραβίαση του κοινοτικού πλαισίου και πώς αντιδρούν οι τελωνιακές αρχές, πώς ορίζεται δηλαδή αυτό το πλαίσιο των παραβιάσεων των κοινοτικών κανόνων. Θα ήθελα να γίνει ένας γύρος των ομιλητών. Η κυρία Γιάκων Σάρη θα μπορέσει να σχολιάσει και θα επανέλθουμε στην Επιτροπή και μετά θα έχουμε σχόλια από την εισηγήτρια. Σόλτες. Είναι εδώ. Τούντα. Σχόλια έχετε. Όχι, όχι. Γιάκων η κυρία Γιάκον μετά θα επανέλθουμε στην Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Επιτροπή για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση και πολύ χρήσιμα παραδείγματα που μας ε, έδωσε έχουν επιλεγεί πολύ σωστά και ε, αυτό επηρεάζει και τις δικές μας θέσεις. Ε, το ΕΛΚ είπε ότι η άποψη του Κοινοβουλίου είναι αρκετά σαφής, αν όχι απόλυτα σαφής σε αυτή την πρώτη συζήτηση. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε την ε, προγενέστερη γνωμοδότηση με μεγάλη πλειοψηφία. και δεν θέλαμε να συμπεριλάβουμε τις εξαγωγές σε αυτή την κεφαλίδα. Το ζήτημα είναι κατά πόσο αυτός είναι ένας σκόπιμος τρόπος προσέγγισης του θέματος που μας απασχολεί. Έγινε μία συνάντηση των σκιωδών και την επόμενη εβδομάδα προβλέπεται τριμερής διάλογος και έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε από πιο κοντά αυτά τα ζητήματα που σχετίζονται με τις εξαγωγές και να βρούμε μία λογική λύση. Όμως, τώρα μπορώ να πω ότι υπάρχουν πολλά διακυβεύματα, όπως η προστασία δεδομένων και η πρόληψη της κακής χρήσης δεδομένων. Θα ήθελα να ακούσω και τις απαντήσεις της Επιτροπής ε, στα ερωτήματα των συναδέλφων. Ωραία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο για να απαντήσει. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο για να απαντήσω στις ερωτήσεις ε, που ετέθησαν και οι συνάδελφοί μου εν συνεχεία μπορούν να συμπληρώσουν ό,τι θα έχω πει. Φυσικά πολύ καλά γνωρίζετε, μάλλον ε, γνωρίζουμε τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πολύ σωστά είπε και η συγκήτρια ότι έχουμε τριμερή διάλογο την επόμενη εβδομάδα. Πρέπει λοιπόν να βρούμε μια λύση για τα ζητήματα επί των οποίων Συμβούλιο και Κοινοβουλίο δεν έχουν την ίδια άποψη. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλουμε κατά κάποιο τρόπο να διευκολύνουμε την επίλυση συμβαστικών, την εξέβριση συμβαστικών λύσεων. Και η σημερινή συνεδρίαση μπορεί να βοηθήσει προς αυτό, να ενημερωθούμε δηλαδή για το τι διακυβεύεται. Έρχομαι στα σχόλια και προσώπου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Στόχος είναι η καταπολέμηση της απάτης ε, και της Όλαφ ε, και ημών και ο κανονισμός 515 αυτό το σκοπό έχει. Δηλαδή να αντιμετωπίσει, να διορθώσει τις παραβιάσεις της τελωνιακής κοινωτικής νομοθεσίας. Θέλω να σας θυμίσω τι έκανε το Συμβούλιο. Συμπεριλαμβάνονται μεν στο κείμενο του Συμβουλίου αυτά τα μηνύματα κατάστασης αμπροματοκιβίων για τις εξαγωγές. Όχι όμως όλα, αλλά κάποιες κατηγορίες αναφέρονται μόνο. Δηλαδή δεν πρόκειται για όλα τα CSM εξαγωγών δεν εμπίπτουν όλα στο πλαίσιο του κανονισμού, παρά μόνο ένας περιορισμένος αριθμός εξ αυτών, τα οποία θεωρούμε ότι διευκολύνουν, ε, θεωρεί το Συμβούλιο, ότι διευκολύνουν την καταπολέμηση της απάτης. Το περιεχόμενο είναι περιορισμένο στο κείμενο του Συμβουλίου. Και οι, ε, κατηγορίες ε, και τα συγκεκριμένα μηνύματα είναι περιορισμένα. Δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες, απλά σα ξεκαθαρίζω ότι το κείμενο του Συμβουλίου δεν καλύπτει όλο τον αριθμό, ούτε όλες τι κατηγορίες ε, των CSM εξαγωγών. Επίσης, αυτά τα CSM, αυτά τα μηνύματα κατάσταση εμπορεύμα το είπε και ο κύριο Ράι, δεν είναι ονομαστικά, δεν περιλαμβάνουν ονομαστικά δεδομένα. Μιλάνε για τι κινήσει ε, των ε, εμπορευματοκιβωτίων. Δεν υπάρχουν ε, ονόματα, δεν υπάρχουν ονομαστικά δεδομένα. Βέβαια, παραδέχομαι ότι αν κάποιο συνδυάσει αυτά τα στοιχεία με τι διασαφήσει, για παράδειγμα, ή με άλλα εξειδικευμένα έγγραφα, τότε βρίσκει τι ονομαστικέ πληροφορίε. Όμω, θεωρούμε ότι προσφέρουμε με το κείμενο επαρκείς ασφαλιστικέ δικλείδε και το είπα και στι εισαγωγικέ μου παρατηρήσει. Υπάρχουν ζητήματα εχεμήθεια, ε, εμπορικών απορρίτων. Αυτά είναι σημαντικά για την Κομισιόν. Τα καταλαβαίνουμε ε, τα επιχειρήματα του Κοινοβουλίου. Καταλαβαίνουμε και την άποψη του κλάδου. Και νομίζω ότι στο κείμενό μας προβλέπουμε αυτές τις ε, ασφαλιστικές δικλείδες. Φυσικά και είμαστε όμως διατεθειμένοι να μελετήσουμε ακόμη περαιτέρω το θέμα και αν βρούμε μια λύση που ε, διευκολύνει, ε, λαμβάνοντας υπόψη και τους κανόνες περί απορρίτου, θα το πράξουμε. Δεν ξέρω αν ο κύριος θέλει να προσθέσει κάτι ο κύριος Ράις. Ένα πρακτικό παράδειγμα θέλω να αναφέρω που δεν σχετίζεται με την αρμοδιότητα της Όλαφ, αλλά παρόλα αυτά δείχνει ότι ο κανονισμός 515 είναι μια δυνατότητα που ανοίγει την πόρτα για έρευνες και ενδεχομένως επιβολή κυρώσεων και από άλλους φορείς. Για παράδειγμα λοιπόν, έχουμε μια απλή περίπτωση λαθρεμπορίων ναρκωτικών παραβιάζει κάποιος την ε, νομοθεσία όταν δεν δηλώνει την εισαγωγή. Δεν έχουμε τον ε, ε, κανονισμό 515 σε αυτή την περίπτωση. Ισχύει νομοθεσία περί ναρκωτικών. Όμως τι θέλουμε να κάνουμε. Πώς θα ξεκινήσουν τα κράτη-μέλη τις έρευνες, πώς θα ενημερωθούν για την απάτη, γιατί η απάτη από το 1997 και μετά, οπότε και δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά ο κανονισμός αυτός, έχει αλλάξει Πρέπει να προσαρμόσουμε τώρα την κατάσταση. Έχουμε όλο και περισσότερο ή σχεδόν μόνο ηλεκτρονικά δεδομένα. Έχουμε ηλεκτρονικέ διασαφήσει, το e-customs. Ε, συνέχεια εξελίσσεται η κατάσταση και πρέπει και εμεί να προοδεύσουμε. Δεν πρέπει να μείνουμε πίσω ούτε και στον αγώνα κατά τη απάτη. Ευχαριστώ. Κυρία Κέπχαρτ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Είχα ζητήσει το λόγο, αλλά δεν ήθελα να μιλήσω πριν την εισηγήτρια, γιατί πιστεύω ότι βασικά εκείνη έχει εδώ την πρωτοκαθεδρία. Ε, σήμερα δεν συζητούμε τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου. Έχουμε σαφή θέση. Και αυτό είναι θέμα της εισηγήτριας αυτή την εντολή και την αποστολή να την υπερασπιστεί απέναντι στο Συμβούλιο και να έχει ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Εγώ δεν θέλω να μπω λοιπόν στην ουσία όλων αυτών, αλλά να πω κάτι άλλο. Ε, που είπε παρόδο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μου έκανε εντύπωση. Όταν ε, μίλησε για τη συζήτηση με την Αυτιλία και το Παγκόσμιο Συμβούλιο, εκεί λέει σαφέστατα επικοδομητικές συζητήσεις. Πολύ ωραία μας τα λέτε. Τι θα πει αυτό. Και σε μια αναφορική πρόταση που είπατε παρόδο ήταν ότι ναι καλά υπάρχουν εκεί κάποια προβλήματα για το να ορίσουμε ποιος θα έχει πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία. Και αυτή η αναφορική δευτερεύουσα πρόταση δεν είναι καθόλου δευτερεύουσα, είναι κύρια. Γιατί ακούσαμε ότι δεν είναι ονομαστική αυτή η πληροφόρηση, ούτε πρόκειται γι' αυτό στην προστασία των δεδομένων δεν μας ενδιαφέρουν τα πρόσωπα μόνο, αλλά και οι κινήσεις των επιχειρήσεων. Δηλαδή αυτό είναι όντω σημαντικό το θέμα. Ποιος έχει πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία. Ποιος μπορεί να τα συλλέξει, να τα συνενώσει με άλλα στοιχεία. Ποιος έχει την άδεια να ανατρέχει σε αυτά πόσο καλά εξασφαλισμένα αυτά τα δεδομένα και πάει λέγοντας. Γιατί ξέρουμε ότι και εκεί υπάρχουν hackers και όπου είναι οικονομικά συμφέροντα υπάρχουν και τα απαραίτητα χρήματα για να πληρώσει κάποιος hackers και τα λοιπά. Αυτά είναι θέματα και ερωτήματα που μας ενδιαφέρουν και σε σχέση με όλα αυτά και θα περίμενα λίγο παραπάνω πληροφόρηση Εκτός από αυτή την υποπρόταση που λέει έχουμε και κάτι προβλήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να απαντήσει αυτό για την προστασία των δεδομένων και ποιος θα έχει πρόσβαση σε αυτά και σε αυτές τις λεπτομέρειες. Äh, äh, Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που εντοπίσατε και σωστό. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Ράις που έκανε και την παρουσίαση να πει περισσότερα. Έχετε απολύτως δίκιο όμως ότι Εκεί ο νομοθέτης, εκατέρωθεν και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, θα πρέπει να το δει πολύ προσεκτικά. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Δεν ξέρω πώς να εξηγήσει περισσότερο, κύριε κύριο So thank you very much. Uh, σας ευχαριστώ πολύ. Οι επικοδομητικές συζητήσεις με τον Παγκόσμιο ε, Οργανισμό Ναυτιλίες αφορά τα εμπορευματοκιβώτητα κυβότια τα οποία περιλαμβάνουν ε, ονομαστικά στοιχεία, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε πώς ε, μεταφέρονται αυτά τα μήνυματα σε σχέση με το στάτους των κοντέινερ. Τα στοιχεία όμως αυτά ε, είναι ευαίσθητα στοιχεία, γι' αυτό και στον κανονισμό θεωρούμε ότι υπάρχουν υψηλές προδιαγραφές για την προστασία των στοιχείων. Όταν μιλάτε για hacker, βεβαίως Υπάρχει κίνδυνος, αλλά ε, αυτό που έχει σημασία είναι να προστατεύσουμε τα στοιχεία και αυτό προσπαθούμε ακριβώς να κάνουμε. Τα στοιχεία CSM τα οποία συζητήσαμε αφορούν στοιχεία τα οποία ε, σχετίζονται με την μεταφορά αυτών των δεδομένων γιατί έχουμε να κάνουμε με ένα 30% των μηνυμάτων στα εμπορευματοκιβώτια τα οποία μπορεί να συμβουλευτεί κανείς στο διαδίκτυο. Ε, ελπίζω να απάντησα στο έτοιμά σας σε σχέση με τα στοιχεία αυτά και την αντιμετώπιση τους 30% των μηνυμάτων από τα εμπορευματοκιβώτια βρίσκονται ήδη στο διαδίκτυο, αλλά 70% όχι. Ένα 30% εντάσσεται στο διαδίκτυο, αναγράφεται στο διαδίκτυο. Ε, έχω, έχουμε και ένα συνάδελφο από το Κοινό Κέντρο Ερευνών που είναι υπεύθυνο ε, για αυτό το project και μπορεί να προσθέσει ε, κάτι για το 30%. Ο κύριος Ζώης, θα ήθελα να ε, σας πω ότι αυτές τις ε, πληροφορίες μπορούν να δεθούν στους πελάτες από ανοιχτές ιστοσελίδες. Δεν πρόκειται για απόρριτα στοιχεία γιατί δεν υπάρχουν ονομαστικά στοιχεία ή αξίες. Άρα για το CSM τα στοιχεία αυτά είναι ανοιχτά και μπορεί κανείς να ζητήσει τα στοιχεία από τις ε, μεταφορικές εταιρείες. Κυρία Κέπχαρτ, απαντά αυτό στην ερώτησή σας. Έχουμε χρόνο, μπορούμε να συνεχίσουμε όσο θέλετε να ρωτάμε. Και πιο ειδικέ ακόμα θέλετε. Χρόνο έχουμε και είναι εδώ και πυρογνώμονε. Καταλάβατε, διαβάσατε την έκφραση του προσώπου μου πάρα πολύ σωστά. Δεν είμαι απολύτω ικανοποιημένη από τις απαντήσεις που έλαβα. Διότι για να δούμε αυτή τη διαφάνεια. με ναι, το πρώτο ή το δεύτερο παράδειγμα, δεν θυμάμαι ποιο ήταν ακριβώς μια στιγμή να το βρω. Ε, ε, λοιπόν, για να το βρω. Εξάγεται λοιπόν μια μεγάλη ποσότητα τσιγάρων και κάπου πάει το κοντέινερ. Και μετά το στέλνουν πίσω. Και άμα θέλω να κάνω λαθρεμπόριο το βάζω σε άλλο κοντέινερ. Δεν θέλει και πολύ μυαλό αυτό. Ούτε και τεράστια ενέργεια για να το κάνεις. Αυτό το CSM το μήνυμα για το καθεστώς για την κατάσταση του, του εμπορευματοκιβωτίου. Θέλουμε εμείς στο Κοινοβούλιο να μιλάμε μια γλώσσα που να καταλαβαίνει και ο κόσμος που μας ακούει στο διαδίκτυο. Κάπου στην αρχή της συζήτησης κάθισα πολύ ώρα να σκεφτώ και να καταλάβω τι είναι αυτό το CSM που μας λέτε. Ωραία, το κατάλαβα. Είναι ε, ε, δεδομένα ε, ότι αυτό είναι το εμπορευματοκιβώτιο, έχει το τάδε νούμερο και τώρα είναι στο χ λιμάνι και μεταφέρεται στο ψ λιμάνι. Και μετά φεύγει από το ψ με άλλο φορτίο και πάει στο Z ας πούμε, εντάξει. Ή ξαναγυρνάει στο Χ. Εμένα τι με βοηθάει αυτή η πληροφορία, εάν δεν συνδέεται και το περιεχόμενο μαζί. Περί αυτού πρόκειται. Αν είναι απλώς λογιστική καταγραφή το όνομα του κοντέινερ, το αριθμός του, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό μπορεί να είναι μέχρι και δημόσιο και ευχαρίστως. Αυτό το κάνουμε και με τα δέματα που στέλνουμε με το ταχυδρομείο που μας δίνουν ένα νούμερο και μπορούμε να το παρακολουθούμε στο διαδίκτυο που βρίσκεται ανα πάσα στιγμή. Το θέμα είναι πώς θα συνδεθεί το περιεχόμενο με τον περιέκτη που είναι το κοντέινερ και έχει το νούμερο αυτό. Και πώς θέλετε να το ελέγξετε αν δεν έχετε αυτή τη σύνδεση. Και αν την έχετε, το φορτίο με το κοντέινερ, πώς το καταγράφετε και ποιος έχει πρόσβαση σε αυτή την πληροφορία η οποία πού συλλέγεται. Και αυτή η συγκέντρωση και ο συνδυασμός των δεδομένων είναι αυτό που χρειάζεστε για να κάνετε τον έλεγχο. Και ποιος παρακαλώ θα έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Αυτό με ενδιαφέρει. Επειδή έχουμε χρόνο, θα δώσω το λόγο για μια τελευταία φορά στην Κομισιόν να απαντήσει και μετά εν τέλει η κυρία εισηγήτρια, εκτός αν υπάρξουν βέβαια στο μεταξύ και άλλε ερωτήσει. Ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω. Και εδώ δίκιο έχετε. Και πολύ σωστά εντοπίζετε το πρόβλημα. Ότι θα πρέπει να κάνουμε καλή δουλειά και να πολεμήσουμε ουσιαστικά την απάτη. Να μπορούμε αυτά τα σύστημα των εξαγωγών να τα συνδέουμε και με τα εξαγωγικά δεδομένα πρέπει να τα βλέπουμε αυτά αλληλένδετα. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή μας έχουμε εισαγάγει ε, γενικές ρυθμίσεις για την προστασία δεδομένων και στον κανονισμό 45 του 2001 παραπέμπουμε και στη συζήτηση με το Συμβούλιο αλλά και στη συζήτηση μαζί σας νομίζω μπορεί κανείς να πει καταλάβαμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερες ασφαλιστικές δικλίδες και μπορώ να σας πω ότι το Συμβούλιο στην πρότασή του που επί της αρχής καταρχήν τα έχει δεχτεί αυτά τα CSM των εξαγωγών έχει και άλλες ε, ρυθμίσεις και διατάξεις εγκρίνει το Συμβούλιο περί ε, εμπορικού απορρίτου. Δεν μπορώ τώρα να σας πω λεπτομέρειες, ε, είναι και θέμα περαιτέρω διαπραγματεύσεων, αλλά και το ίδιο το Συμβούλιο έχει συμπεριλάβει βρίες διατάξεις για την προστασία του εμπορικού απορρίτου. Προηγουμένως αναφέρθηκε γι' αυτό πώς κινούνται οι εμπορικές ροές των επιχειρήσεων και κατά πόσο αυτό είναι θέμα που πρέπει να προστατεύεται και αν θα έχουν πρόσβαση στα κράτη-μέλη ή αν θα περιορίζεται αυτό σε κάποιες υποθέσεις που αφορούν μόνο το ίδιο το κράτος ή αν είναι γενικότερα. Δεν μπορώ δυστυχώς να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες τώρα, διότι έχουμε την αρχική μας θέση στην Κομισιόν, αλλά πώς να πω, εγώ είμαι πρόθυμη και ακούω με μεγάλη προσοχή αυτά που λέτε για το θέμα, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε μια λύση. για να εξασφαλίσουμε και την προστασία των δεδομένων και την προστασία του εμπορικού απορρίτου. Okay, mein Kollege hat mir gerade noch eine... Μου δίδει η συνάδελφος τώρα ένα με εδώ ε, του συναδέλφου από το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο. Δεν ξέρω, θέλετε να πείτε κάτι συμπληρωματικά, κύριε Ζωή, παρακαλώ. Σε σχέση με αυτά που μόλις είπα. Έτσι κατάλαβα καλά. Uh, uh, θα ήθελα να προσθέσω ότι τα κράτη-μέλη και οι τελωνιακές αρχές έχουν ε, πρόσβαση στα ονομαστικά στοιχεία, γιατί ε, έχουν ήδη πρόσβαση για την δικά τους στοιχεία. Και δεν θα αλλάξει η κατάσταση ως προς την τρέχουσα. Εισηγήτρια, σας ευχαριστώ πολύ για τις ε, πληροφορίες αυτές που πιστεύω ότι θα μας κάνουν ε, να σκεφτούμε και όλες αυτές τις νέες παραμέτρους. Όταν έγινε αποδεκτή αυτή η πρόταση σε πρώτη ανάγνωση με τόσο μεγάλη πλειοψηφία, είχα σκεφτεί ότι δεν θα δημιουργήσει και μεγάλα προβλήματα. Να που προέκυψαν όμως και παρόλα αυτά τα έχουμε όλα μελετήσει πάρα πολύ προσεκτικά και όπως σας είπα έχουμε αύριο συνάντηση με τους κοιόδης εισηγητές και την επόμενη εβδομάδα ξεκινάμε με τον τριμερή διάλογο.